Okay, colleagues, can I bring the meeting to, to order? This may... Αγαπητοί συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε. Μπορεί να μην σας ξαφνιάσω, να σας ξαφνιάσω, αλλά δεν έχουμε πίεση χρόνου σήμερα. Η μόνη πίεση που έχουμε είναι να μείνουμε μέσα στην αίθουσα τόσο ώστε να φτάσει ο καφές και το τσάι. Πράγμα πολύ σημαντικό, όπως λέει και ο Πέτερ. Και έτσι περνάω στι ανακοινώσει του Πρόεδρου καταρχάς, αποφάσεις της συνεδριάσεως των συντονιστών 14 και 25 Νοεμβρίου. Δύο συνεδριάσεις. Στις 14 Νοεμβρίου η πρόταση για κανονισμό προσαρμογή στο άρθρο 19.291 της Συνθήκης Λισαβόνας ε, των νομικών πράξεων που έχουν να κάνουν με τις ε, πράξεις ε, εποπτείας οι μόνιμοι εισηγητές για την επιτροπολογία, Κούν και Αλκαντράου, αποφασίστηκε ότι θα αναλάβουν και αυτές τις ε, εκθέσεις. Για, τις, ε, για την αεροπορία, για την πολιτική αεροπορία αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή στο Συμβούλιο ε, όπου θα λέγεται ότι συμφωνούμε να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις για την πρόταση, για την χορύπανση, εφόσον το Συμβούλιο είναι δετεθειμένο να συζητήσει και τα δικαιώματα των επιβατών, για ε, Επίσης ε, λάβαμε γνώση των ε, επιστολών υπαριθμών 26 της 4ης Νοεμβρίου και 27 της 11ης Νοεμβρίου και αν χρειαστεί υποχωρήπαν στην αρχή να συζητείτε την επόμενη συνεδρίαση. Για τους συντονιστές της χθεσινής ημέρας έγινε παρουσίαση από την μονάδα για την ασφάλεια ε, στις ε, αεροπορικές μεταφορές όσον αφορά την απαγόρευση, το λεγόμενο μαύρο, τη μαύρη λίστα, την απαγόρευση πτήσης. Ε, ο Πρόεδρος υπενθύμησε ότι αν δεν εγερθούν μέχρι τις 29 Νοεμβρίου τη μέρα Παρασκευή θα αποσταλεί η σχετική επιστολή στην Επιτροπή για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης των Πολιτειών για τους μόνιμους συγητές μεταφορών και τουρισμού. Θα έχουμε πάλι τον μόνιμο μας ηγητή για την επιτροπολογία. Ε, λάβαμε γνώση της επιστολής 28 μια νέα έκδοση προς την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων για τις ε, προτάσεις όμνιμπους που θα ευθυγραμμίζουν την νομοθεσία με τη συνθήκη της Λισαβόνα σχόλια έως τις 29 Νοεμβρίου το μεσημέρι, μερα Παρασκευή, στα διάφορα συζήτηση για τη στάση δεύτερη ανάγνωση του ταχογράφου. Αυτά. Είπαν οι συντονιστές. Είστε όλοι ευχαριστημένοι. Πολύ καλά. Ένα λεπτάκι να βουτήξω και το φακελάκι του τσαγιού και να προχωρήσουμε στην έκθεση του κύριου Φιντάτσα και του ψηφορία. ανάπτυξη υποδομών ελεκτικών καυσίμων. Έχετε, λάβει, έχετε όλες τις κάρτες μαζί σας. Θα κάνουμε πρώτα μία δοκιμή παρακαλώ. Δοκιμαστική ψηφοφορία, να επαληθεύσουμε πώς είναι και από το ΕΛΚ. Ψήφισαν όλοι. Είστε σίγουροι. Φαίνεται να έχουν ψηφίσει όλοι πια. Πέρα τη ψηφοφορία. και συγχαρητήρια. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είναι υπεράριθμο για μια φορά σήμερα. Συγχαρητήρια. Να, που καταφέρει ο Ματσίρ επιβάλλει και την πειθαρχία του στο ΕΛΚ. Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Έχουμε τις τροπολογίες 73 και 74. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 1. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μου αρέσουν αυτές οι ψηφοφορίες. Συμβασμός 5, υπέρ. Κατά εποχές συγκρίνεται. Συμβασμός 6 υπέρ. Κατά. Εποχές συγκρίνεται. Πάμε στο 6 α νέο Τροπολογία 3.42 και τροπολογία 42. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 3.41. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 55, 342, τμήμα 2, 56, 62, 72, όλα μαζί. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 343 Τέιλορ. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 38 ως προσθήκη. Υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 59-60-61 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 344 υπέρ. Κατά εποχές. Νομίζω απορρίπτεται να ελέγξουμε όμως. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Κατόπιν γλωσσική τροποποίηση, μετά πάμε στο 345 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 63 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3, 6 υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στη 41, γιατί οι υπόλοιπε καταπίπτουν. 41 ήτρε, υπέρ. Κατά. εποχές, απορρίπτεται. 65 και 347 ταυτόσημες, υπέρ. Κατά. εποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται 350 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για την επόμενη υπέρ κατά αποχές για την 351 να ελέγξουμε άρχεται ψηφοφορία ψηφίζετε όλοι πέρας εγκρίνεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 353 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Παραρτήματα τώρα. Συμβιβασμό 7. Υπέρ. Κατά. εποχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβασμό 8. Υπέρ. Κατά. εποχέ Εγκρίνεται. Συμβασμός 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντας. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 77 Τέιλορ, υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 11 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 12. Συμβιβασμός 12 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τέσσερα του ηγητή υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 13 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Δέκα του ηγητή υπέρ. Κατά εποχές Νομίζω εγκρίνεται να ελέγξουμε. Άρχεται ψηφοφορία για την τροπολογία 10. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στην 94 της κυρίας Μπιλμπάου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 πίπτη 11 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 97 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 98 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται Συμβεσμό 14 υπέρ κατά Αποχέ εγκρίνεται 13 του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 15 υπέρ κατά εγκρίνεται. Για το κύριο Τριγκάντα 1,7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16, συμβιβασμός 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμό 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 κυρίες Μπιμπάου υπέρ κατά Κατά. εγκρίνεται 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται. 141 υπέρ κατά εποχές συγκρίνεται. 142 υπέρ κατά να ελέγξουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 45, πέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 144 προσθήκη, υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 25, εισηγητή, υπέρ. Κατά. Εποχές Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα την πρόταση που στροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 30 υπέρ, 7 κατά. Καμία αποχή. Εγκρίνεται. Το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα. Τρίτη πέρα από τα κατά. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στον κύριο Φιντάντσα. Περνάμε τώρα στην ε, ψηφοφορία σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Άρχεται η ψηφοφορία. Τις διαπραγματεύσεις. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα. 37 κατά καμία αποχή. Σας ευχαριστώ. Και ολοκληρώνουμε τη σημερινή συνεδρίαση του πρωινού. Να σας υπενθυμίσω κυρίες και κύριοι ότι, αυτό το, ότι σήμερα το απόγευμα πριν να φύγετε όλοι Έχουμε ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Μπρένερ από τη Eurocontrol και κατόπιν με τους τέσσερις συντονιστές. Προσπάθησα να τους επισημάνω ότι έχουμε χρονικούς περιορισμούς και κατόπιν ε, έχουμε τις λιμενικές υπηρεσίες. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να επανέλθετε στις 3 για να ξεκινήσουμε έγκαιρα. Γιατί θα ήταν πολύ άσχημο να είναι άδεια η αίθουσα. Και επίσης να σας πω ότι για τους σκιώδεις, για το πακέτο των σιδηροδρόμων, έχετε τώρα την αίθουσα στη διάθεσή σας, αν θέλετε να κάνετε κάποια δουλειά σε σχέση με αυτό. Αλλά οι θα τα πούμε το απόγευμα.